Ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στην ε, έγκριση των πρακτικών της συνόδου, της περίοδου συνόδου της 8 Οκτωβρίου του 2009. Πρακτικά και κείμενα που υιοθετήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου είναι στη θέση σας ήδη και ρωτώ αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να στέκανε το λόγο. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Ενημερώσει. Ανακοινώσει. Οι κύριοι